Καλημέρα σας συνάδελφοι. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να αναφερθώ στο γεγονός ότι σήμερα έχουμε την επέτειο ενός τραγικού γεγονότος. Πριν από 20 χρόνια, στις 23 Μαΐου, ο δικαστής Τζοβάνι Φαλκόνε, ε, που πολεμούσε τη μαφία, η σύζυγός του, Φραντσέσκα Μορβίλο, και οι σωματοφύλακες Βίτο Σκυφάνη, Ρόκο Ντιτσίλο και Αντώνιο Μοντινάρο ε, σφαγιάστηκαν στο Καπάτσι. Σήμερα ε, έγινε μία τελετή στο Παλέρμο για τα θύματα της μαφία με παρουσία του Προέδρου Τζόρτζο Ναπολιτάνο και του Πρωθυπουργού Μαριο Μόντι. Θα ήθελα να καλέσω το Σώμα να συμμετάσχει στην επέτειο αυτή ε, τιμώντας το παράδειγμα και την αφοσίωση του δικαστή Φαλκόνε και να τιμήσει τη μνήμη όλων εκείνων που πέθαναν στον αγώνα για την ε, αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Ενός λεπτού σιγή παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι όλοι έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες για τις ψηφοφορίες. Δεν είναι μακρά η ψηφοφορία σήμερα. Ελπίζω να προχωρήσουμε γρήγορα. Πολλοί συνάδελφοι γνωρίζω ότι θέλουν να φύγουν για να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν την Οικονομική Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Ο κύριος Μποστινάρου παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, προχθές στην Αλβανία έγινε μια μεγάλη καταστροφή ε, τροχαίο με 14 νεκρούς ένα λεωφορείο ε, έπεσε σε χαράδρα, 14 ε, άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και την συμπάθειά μας προς τις οικογένειες των θυμάτων και τραυματισθέντων. Ταυτόχρονα θα ήθελα να εκφράσουμε και, μια, και την αλληλεγγύη μας ε, με τη προς αλβανικό λαό. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου που θέσατε το ζήτημα αυτό το οποίο καταγράψαμε και εκφράζει ε, κάθε ε, συμπάθεια το Κοινοβούλιο προς τα θύματα του ατυχήματος αυτού. Ε, θα ήθελα επίσης να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς όλους τους φυλακισμένους μετά από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Τώρα, έκθεση Ραούλ Ρωμέβα Ιερουέδα, αποκατάσταση του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και την Μεσόγειο. Ε, το η πρώτη ενότητα σε ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Πρόταση της Επιτροπής ως ετροποποιήθη. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μετά την παράγραφο 1 υπάρχει η τροπολογία 4 της Επιτροπής Αλίας τίθεται σε ψηφοφορία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Να το ελέγξουμε αν θέλετε. Ε, αρχίζει η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 4. Ε, πέρας της ψηφοφορίας δεκτή. Τώρα, το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος ε, τίθεται σε ψηφοφορία, συνολικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή με πολύ ισχυρή πλειοψηφία συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ο εισηγητής παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την υποστήριξη στην έκθεση και βεβαίως έπαιξε ε, ρόλο ο κύριος Βάτσον ε, ε, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθούμε σε εκείνο ε, και είναι πολύ σημαντικό να ζητήσουμε να μην εκδοθεί στην Κωνσταντίνα. Ε, η επόμενη έκθεση είναι του κυρίου Ρικέ. Απαιτήσει διπλού κήτου ή ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κήτου. Ε, πρώτη ενότητα τη ψηφοφορία. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα, η πρόταση τη Επιτροπής, η τίθεται ψηφοφορία όσο τροποποιήθηκε υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Και τώρα η πρόταση νομοθετικού ψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Έγινε δεκτή συγχαρητήρια κύριε Ρικέ. Η έκθεση Γκαρθία Χέρο Καραμπάλο αλληλευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται συμφωνίες, στη Συμφωνία Αλληλευτικής σύμπραξη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας τη Μοζαμπίκη. Τίθεται σε ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορία. Και αυτό έγινε δεκτό. Συγχαρητήρια κυρία Χερό Καραμπάλο. Και περνάμε στην έκθεση της κυρίας Ποδήματα για ένα κοινό σύστημα φόρου και των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και η πρώτη είναι η τροπολογία 40. Ονομα, ε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 32 τροπολογίες από την Οικονομική Επιτροπή. Ψηφίζομαι όλες μαζί υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. Ψηφίζομαι την τροπολογία 11, τμήματική ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα της 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Να ελέγξουμε. Ελέγχομαι ηλεκτρονικά τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας του ηλεκτρονικού ελέγχου. Δεκτή. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 52, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Προχωρούμε στην τροπολογία 38, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας Απερίφθη 37 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 43 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κατέπεσε η 42, συγγνώμη. 43 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 41, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τώρα, η πρόταση της Επιτροπής ως ετροποποιηθεί. πέρ. Κατά. Δεκτή. Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτώ με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία Ποδηματά. Τώρα έκθεση της κυρίας Δεσσαρνές για την ανισορροπία στο εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα διορθωτικό σε όλες τις γλωσσικές εκδοχές της έκθεσης. Η λέξη «άιλη» έχει αντικατασταθεί από την πνευματική. Για ορισμένους μπορεί να σημαίνει το ίδιο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι το ταυτόσιμη. Η τροπολογία υπαριθμών ένα ψήφι Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και ερχόμαστε στην παράγραφο 1. Έχουμε κατά τμήματα ψηφοφορίες. Όχι, χωριστές. Παράγραφος 3 πρώτα. Όχι, παράγραφος 1, διορθώνει ο πρόεδρος. Παράγραφος 1, ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο, ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 11, σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο, ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σε δύο τμήματα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 15 σε δύο τμήματα. Ψήφι υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Σε δύο τμήματα. Υπέρ. Του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το, παράγραφος 29, δύο τμήματα, τμήμα πρώτο, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 30. Σε δύο τμήματα και πάλι, τμήμα πρώτο ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα, νομαστική κλίση, ανοίγει τώρα. The Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Παράγραφος 37. Δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη και η λατινικό. Υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για την αιτιολογική σκέψη και η τώρα. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η αιτιολογική σκέψη την λατινικό σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στο σχέδιο ψηφίσματος στο σύνολό του. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Ντεσανέζ. Το Επόμενο θέμα, η έκθεση David Martin, δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ενημερώσω το, το Κοινοβούλιο, οι τροπολογίε 1 και 3 έχουν αποσυρθεί και η, τροπολογία 31 κηρύχθηκε μη παραδεκτή. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στην τροπολογία 18, ψήφι υπέρ. Α, συγγνώμη, έχασα μια σελίδα, λέει ο πρόεδρο. 19 τροπολογίε 4 πολιτικών ομάδων. Ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τώρα έχουμε τη 18 ψήφι ΠΕ. Α, συγγνώμη, είναι ονομαστική εκκλήση, λέει ο Πρόεδρος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 19 και πάλι ονομαστική, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρες, Εγκρίνεται. 22. Ορίστε. Η κυρία Ντεκεζέ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Μπορείτε λίγο να σταματήσετε 30 δευτερόλεπτα για να συνεννοηθούμε. Δεν έχουμε καθόλου τον ίδιο κατάλογο ψηφοφορίας και δημιουργούνται προβλήματα. Um, Can someone help Mrs. De Kaiser with the voting list? Mrs. Harms. Κυρία Χάρμς, εσείς τι λέτε. Perhaps the um, socialist group could follow Mr. Martin. Οι σοσιαλιστές μήπως να ακολουθούν τον κύριο David Martin.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 Έρχεται ένα οσίες ε, του κυρίου Ολάντ να σα βοηθήσει. Yeah, yeah. Has he got it? Okay. Ah, Steve Hughes is in charge. Ah, Steve Hughes ε, είναι υπεύθυνο. ωραία. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Στροπολογία 22. Είστε σίγουροι πώς θα ψηφίσετε γιατί είναι και ονομαστική, έτσι. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία επαριθμών 22. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στην τροπολογία παρφών 5. Ψήφι πέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία. Έλεγχο θέλετε. Ας το ελέγξουμε. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την τροπολογική περιφέρον 5. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Όντως απερίφθη. Και ερχόμαστε στην αντίστοιχη παράγραφο της τροπολογίας 12. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6, those in η έξι ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η αντίστοιχη παράγραφος στι τροπολογίε 12 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα. Μετά την παράγραφο 7 έχουμε στο άρθρο 7, συγγνώμη, μετά την παράγραφο 2 ψηφίζουμε τη 12, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 15, ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 ψήφι κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα η πρόταση όπως τροποποιήθηκε ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Και ο κύριος Μάρτιν έχει το λόγο. Θέλει κανείς να στήσει αναβολή της τελικής ψηφοφορίας. Ναι, Πρόεδρε για να έχουμε περαιτέρω συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να προτείνω αναβολή της τελικής ψηφοφορίας για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος και ελπίζω να το δεχτείτε. Έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο ε, μέχρι σήμερα και σήμερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πιστεύω ότι θα πρέπει τα τρία θεσμικά όργανα να συνέλθουν και να συμφωνήσουν για αυτό το θέμα. Ένα ομιλητή υπέρ. Υπάρχει κατά. Ψηφίζουμε. Υπέρ της πρότασης του κύριου Μάρτιν. Κατά της πρότασης του κύριου Μάρτιν. Αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Ευχαριστώ όλους σας. Καλή σας όρεξη. the